κοινωνία των πολιτών μπορούν να αντλήσουν κονδύλια από εκεί για να ε, καταπολεμούν στην πράξη τέτοιε διακρίσεις. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ σας ευχαριστώ κυρία Πίτροπε, κυρία Χέντεγκαρτ. Έχω λάβει έξι ψηφίσματα από έξι πολιτικές ομάδες, ε, συντηρητικοί, ΕΛΚ, πράσινοι, φιλελεύθεροι, σοσιαλιστές και δημοκράτες. Και εδώ ολοκληρώνεται η συζήτηση και εγώ. Ε και η ψηφοφορία θα γίνει στη συνέχεια. Επόμενο θέμα. Ελευθερία τη έκφρασης στη Λευκορωσία, ιδιαίτερα η υπόθεση του Αντρέη Πότσομπουτ. Θα δώσω το λόγο στου συντάκτε πρώτα ο κύριος Κάτσμαρεκ για ένα λεπτό. Επίτροπε κυρίε και κύριοι, Είμαι ικανοποιημένος που μπορώ να πω ότι ο κύριος ε, Ποσκομπούτ ε, απελευθερώθηκε, αποφυλακίστηκε, αλλά το ζήτημα δεν έχει ακόμα κλείσει, διότι ό,τι συμβαίνει στην Λευκορωσία είναι πολιτικής φύσης και ε, ο νόμος ε, και οι σχετικές διατάξεις χρησιμοποιούνται προκειμένου να διώκονται οι ακτιβιστές ε, για τα ανθρώπινα δικαιώματα. Θα πρέπει λοιπόν εμείς όπως πάντα να υπερασπιστούμε τις ελευθερίες της έκφρασης. Η ελευθερία της έκφρασης παραβιάζεται καθημερινά στην Λευκορωσία και ο κύριος Πόσκομπούτ διώκεται και διώχθη για αυτόν τον λόγο. Πρέπει να απελευθερωθούν όλοι οι κρατούμενοι για παρόμοια δικήματα. Ευχαριστώ. Και τώρα η κυρία Λούνατσεκ, παρακαλώ. Για ένα λεπτό. Α, Πρόεδρε, επιτροπές στα Αγγλικά, η κυρία Λούνατσεκ, κυρίες και κύριοι. Και εμεί εξεπλάγημεν ευχάριστα κατά κάποιο τρόπο από το γεγονό ότι τον απελευθέρωσαν το περασμένο Σάββατο τον κύριο Πότσοβουτ. Όπω είπε όμω ο προλαλή σα. Ε, δεν μπορούμε να καθησυχάζουμε ούτε να μα ε, ικανοποιεί η κατάσταση. Ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά τα δικαιώματα ε, της αντιπολίτευσης των δικηγόρων, των δημοσιογράφων και άλλων ακτιβιστών στη Λευκορωσία. Ακούστηκαν επικρίσεις για τον ε, τρόπο με τον οποίο κυβερνάει ο κύριο Λουκατσέγκο. Είναι σχεδόν δικτατορία. Ε, είναι όμω τελευταία δικτατορία που παραμένει στην Ευρώπη και έχουμε ξαναπεί και χαίρομαι που το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είναι ενωμένο απέναντι σε οποιαδήποτε ε, παραβίαση ε, ελευθερίας έκφρασης σε ευρωπαϊκή χώρα. Στο ψήφισμά μας λοιπόν ε, απαιτούμε από τις αρχές της χώρας να σταματήσουν κάθε πίεση και κάθε καταπίεση και καταστολή απέναντι σε δημοσιογράφους, ακτιβιστές, ε, ε, αντιφρονούντες και να αφαιθούν ελεύθεροι όλοι οι πολιτικοί κρατούμενοι. Εδώ πέρα είναι Ευρώπη και η Λευκορωσία είναι ευρωπαϊκή χώρα. Δεν έχουν ε, θέση στην Ευρώπη τέτοιες συμπεριφορές. Ευχαριστώ κυρία Λούνατσεκ. Η κυρία Σάκη για δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε τη συνάλφη. Μπορεί να απελευθερώθηκε ο κύριος ε, Πότσο που τα λέξη ακολουθεί να αντιμετωπίζει ε, τις κατηγορίες αυτές, δηλαδή για τις δραστηριότητες του ως ακτιβιστή και ως μέλος μιας ε, πολωνικής μειονότητας. Δεν είναι ο μόνος δυστυχώς η κατάσταση με τους περμάξεων των δικαιωμάτων που εκπροσωπούν την κοινότητα των πολιτών, δημοσιογράφοι ε, και η κατάσταση των ε, των πολιτών στη Λευκορωσία επιδεινώνεται. Η ελευθερία έκφραση και online στο διαδίκτυο ε, είναι αντικείμενο καταστολή πιέσεων και αυτό γίνεται μάλιστα με την ίδια την βοήθεια εταιριών Ευρωπαϊκής Ένωσης που δίνουν στη Λευκορωσία τη σχετική τεχνολογία που τη επιτρέπει να προβαίνει σε αυτή την καταστολή. Έχουμε λοιπόν κατάφαση παραβίαση ανθρωπίνων δικαιωμάτων και με τη βοήθεια τεχνολογία ευρωπαϊκής. Αυτό πρέπει να τερματιστεί. Είναι η Λευκορωσία η τελευταία δικτατορία στην Ευρώπη. Πρέπει το συντομότερο δυνατόν η χώρα να εκδημοκρατιστεί. Η Ευρωπαϊκή Ένωση θα πρέπει να στείλει ένα ξεκάθαρο μήνυμα στις αρχές της Λευκορωσίας ότι ε, δεν ε, είναι καλοδεχούμενες ε, στην συνεδρίαση της Γιούρνη το τέλο του μήνα αυτού. Υπάρχουν όροι και πρέπει να τηρηθούν. Είναι αυστηρή η όρη αυτή. Οι αρχέ τη Λευκορωσία πρέπει να δεσμευτούν, να σέβονται το κράτο δικαίου, να σέβονται τα ανθρώπινα δικαιώματα. Κάτι άλλο στο που έχουν δηλώσει και οι ίδιοι ε, το 2009 στην ε, διάσκεψη κορυφή. Θα πρέπει όμως ε, ταυτόχρονα να κλιμακώσουμε τις επαφές μας με τις ε, ανθρωπικές οργανώσεις στη χώρα, με, τους, με την κοινωνία των πολιτών ο περιορισμό τη ελευθερία του τη συνεταιρίζεσαι, τη ελευθερία έκφραση, όλα αυτά πρέπει να έρθουν. Ο σεβασμό αυτών των ελευθεριών είναι βασικό ακρογωνίο λίθο τη δημοκρατία που ε, ότι η ηρωνία ε, είναι κάτι για το οποίο έχουν δεσμευτεί οι λευκορωσικέ αρχέ και έχουν πει ότι θα σέβονται αυτές τις ελευθερίες. Ε, θα πρέπει λοιπόν να επιβάλλουμε επιπλέον κυρώσει και να κλιμακώσουμε τι προσπάθειε μα ώστε να μην παραμείνουν μόνο στα χαρτιά όλε αυτέ οι δεσμεύσει των λευκορωσικών αρχών. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ρέπο, για μισή λεπτό. Κύριε Πρόεδρε, ο Ανδρέ Πρέτσοβούτ ε, είναι δημοσιογράφος πολωνικής καταγωγής και εκπροσωπεί μειονότητα. Ήταν στη φυλακή και περίμενε ε, να γίνει ε, δίκη του. Ένας ε, δημοσιογράφος που εκφέρει άποψη για το πρόσωπο του κυρίου Λουκασέγκο στη Λευκορωσία για την κοινωνική κατάσταση καταλήγει στη φυλακή. Η πένα έχει μεγάλη εξουσία και όταν κάποιος γράφει κάτι μπορεί να βρεθεί στη φυλακή για χρόνια, πολλά. Αυτό έχει να κάνει με τον εγωισμό του Προέδρου Λουκασέγκο και με τις αδυναμίες του δεν υπάρχει δημοκρατία, δεν υπάρχει κοινωνία των πολιτών και δεν του αρέσουν όλα αυτά. Γιατί αυτά σημαίνουν ότι ε, έτσι λύγει η δική του εξουσία. Ε, ε, βέβαια έχει αφαιθεί ελεύθερο στο μεταξύ ο κύριος ε, Πότσοβουτ, πολύ καλή είδηση αυτή, χάρη στην πίεση και την άμεση κριτική, χάρη στο διαδίκτυο και χάρη στην άμεση δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Κοινοβουλίου. Η Διεθνής Αμνηστία ήδη τον είχε ε, χρήση πολιτικό κρατούμενο και κρατούμενο λόγω της ελευθερίας της έκφρασης. Είναι και άλλοι κρατούμενοι όμως και περιμένουν να φεθούν ελεύθεροι. Η φυλάκιση κάποιου λόγω των πεπιθήσεων του συνιστά ε, κατάφορη παραβίαση των θεμελιωδών ε, και παγκοσμίων δικαιωμάτων και παραβιάζει και το Σύνταγμα της Λευκορωσίας. Το, η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και τέλη του μηνό θα πρέπει να εξετάσει περισσότερο και σε μεγαλύτερο βάθο την κατάσταση στη Λευκορωσία. Ευχαριστώ κύριε Ρέπο. Ο κύριο Μαστάλκα, για ένα λεπτό. Πρόεδρε, θα ήθελα και εγώ να συμφωνήσω με εκείνου που σήμερα υπερασπίζονται ε, τους ε, κρατουμένου συνείδησης. Καθένας θα πρέπει να έχει το δικαίωμα να εκφράσει την άποψή του και να μην διώκεται. Αλλιώς πρέπει να το προστατεύουμε. Αλλά είμαστε επιλεκτικοί ε, στην προσέγγιση μας. Γιατί έχουμε τέτοια επιλεκτικότητα και ε, περνάμε τέτοια ψηφίσματα που οδηγούν σε διχασμό και σε αντιπαράθεση με χώρες. Σήμερα συζητούμε για τον Ανδρέη Ποτσομπούτο, αλλά φοβούμε ότι δεν πρόκειται να ενδιαφερθούν για άλλους αντιφρονούντες όπως τον Τζούλια Ασάνς αυτός που αποκάλυψε τα βρώμικα μυστικά ε, διαφόρων τώρα μπορεί να διώκεται ευχαριστώ κύριε Μαστάλκα τελευταίο συντάκτης Κύριε Πόσελτ, έχετε γαλάζια κάρτα. Κύριε Μαστάλκα, επιτρέπετε ενδιάμεση ερώτηση του κυρίου Πόσελτ. Θέλω να ρωτήσω τον κύριο Μαστάλκα. Ο πρέσβης της Λευκορωσίας στην Πράγα επένεσε τα μάλα και ευχαρίστησε τον πρόεδρο Κλάους για την επικοδομητική του στάση απέναντι στη Λευκορωσία. Και θέλω να ρωτήσω τον κύριο Μαστάλκα πώς το αξιολογεί. Ε, κύριε Μαστάλκα, ε, κύριε ε, Πόσελτ, σας ευχαριστώ, αλλά εγώ δεν είμαι εκπρόσωπος τύπου του Προέδρου Κλάους. Ευχαριστώ κύριε Μαστάλκα. Ο κύριος Μικάλσκι, τελευταίο συντάκτης, είπαμε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι. Ε, η κυρία Σάκα είχε δίκιο όταν είπε πως ο κύριο Ποσκομπούτ ε, αποφυλακίστηκε αλλά συνεχίζει να επιγράμματα επί της κεφαλής του η ποινή των 7 ετών δεν έχει ακόμα αθωωθεί. Μην ξεχνάτε ότι μιλάμε για την τελευταία δικτατορία στην Ευρώπη. Γιατί ο κύριος Πότσκομπούτ βρίσκεται στη φυλακή, διότι είναι Πολωνό, είναι αντικαθεστατικός και δημοσιογράφο. Αλλά και όχι μόνο, είναι ένα πολύ καλό, <laughs> Πολωνό, πολύ καλό δημοσιογράφο και πολύ καλό αντικαθεστατικός. Και αυτό παραπήγαινε για τον πρόεδρο Λουκασέγκο. Δεν μπορούσε να το ανεχθεί. Γιατί κατηγορείται, κατηγορείται διότι κάνει καλά τη δουλειά του. Αλλά ε, το ζήτημα είναι εμείς κάνουμε αρκετά. Διότι πάντα θα υπάρχουν κάποιοι σε αυτήν την αίθουσα που δεν θέλουν να κρατούν μια σταθερή και δίκαιη στάση και συμπεριφορά. Το πρόβλημα είναι πως ε, επανειλημμένα έχουμε αποτύχει στο να διατηρήσουμε μια σταθερή γραμμή για αντιμετώπιση του καθόλου της Λευκορωσίας. Ευχαριστώ. Μέχρι εδώ ήταν οι συντάκτε και τώρα οι υπόλοιποι ομιλητέ εξ ονόματο των πολιτικών ομάδων. Ο κύριο Σιλβέστρη πρώτο, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Για νιωστή φορά βρισκόμαστε εδώ για να καταγγείλουμε την έλλειψη ελευθερίας έκφρασης στην ε, Λευκορωσία, με την οποία έχουμε ε, σχέσεις γειτονίας. Ε, ο Ανδρέη Πότσομπουτ ε, φυλακίστηκε διότι επέκρινε τον πρόεδρο Λουκασέγκο. Δεν είναι η πρώτη φορά που καταλήγει στην φυλακή επειδή δυσφήμισε τον πρόεδρο. Είχε καταδικαστεί και πέρυσι για τρία χρόνια διότι επέκρινε τον πρόεδρο από τις στήλες εφημερίδες του. Η ε, ελευθερία έκφρασης ε, και η ελευθερία συνέρχεστε έχουν περιοριστεί και οι ειρηνιστέ έχουν συλληφθεί και καταδικαστεί μετά από συνοπτικές δίκες. Ε, τα άτομα τα οποία έχουν φυλακιστεί για λόγους συνείδησης, ε, για αντιρρησή συνείδησης, ε, του χάνουν κακομεταχείριση στις φυλακές. Όλα αυτά λοιπόν θα πρέπει να τα λάβουμε υπόψη όταν πρόκειται να εξετάσουμε το ζήτημα της περαιτέρω διεύρυνσης της Ευρώπης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκέριγκερ Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η λογοκρισία του τύπου περιορισμό τη ελευθερία έκφραση είναι κοινή πρακτική στη Λευκορωσία. Ο νόμο που έχει επιβληθεί το 2008 και μετά επιτρέπει ξεκάθαρα αυτέ τι πρακτικέ. Το 2011, 95 τουλάχιστον δημοσιογράφοι ήταν υποκαθιστώ επιτήρηση και 30 εξ αυτών ε, φυλακίστηκαν. Ε, στις 21 Ιουνίου ο Αντρέι Πότσομπουτ συνελήφθη. Πρόκειται για δημοσιογράφο και μέλος ε, της Ένωσης Πολωνών της Λευκορωσίας. Κατηγορήθηκε ότι ε, δυσφημεί, ότι λιβελογραφεί κατά του Προέδρου. Έχει μεν απελευθερωθεί, αλλά δεν έχουν, πέσει, δεν έχουν αρθεί και ακυρωθεί οι καταγγελίες ε, που τον βαρύνουν, κατηγορίες. Θα πρέπει να αρχίσει πλέον ε, η Λευκορωσία να τηρεί το άρθρο 24 του συντάγματος ε, που εγγυάται την ελευθερία έκταση στους πολίτες της χώρας. Ευχαριστώ πολύ κυρία Γκέριγκερ. Ο κύριος Τάνοκ. Κύριε Πρόεδρε, η περίπτωση του δημοσιογράφου και ακτιβιστή Ανδρέη Πόρζομπουτ που είναι της πολωνικής μειονότητας στη Λευκορωσία δείχνει την ομότητα και την παράνοια του καθεστώτος του Μίνσκ. Υποτίθεται για τη συκοβατική δυσφήμιση τον συνέλαβε μυστική υπηρεσία για την εφημερίδα του. Στην ε- Ευρωπαϊκή Ένωση ε, είναι θεμητό να ε, επικρίνει την κυβέρνησή σου και είναι και στο δημοκρατικό παιχνίδι. Στη Λευκορωσία όμως αυτή η ελευθερία της έκφρασης τον έστειλε στη φυλακή για τρία χρόνια και κατοίκον περιορισμό ε, μέχρι τη ε, δίκη. Δεν υπάρχει κράτος δικαίου, ούτε ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, ούτε κατά στοιχειώδη ανθρώπινα δικαιώματα. Θα πρέπει να αυξήσουμε τις κυρώσεις μας μέχρι να παραιτηθεί ο Λουκασέγκο και να αποφασίσει ο λαός δημοκρατικά ε, για τους μελλοντικούς ηγέτες. Φτάνει πια στο Κοινοβούλιο. Δεν θέλουμε κι άλλη κούβα στην Ευρώπη. Ε, ευχαριστώ κύριε Τάνοκ. Ο κύριος Μέρφυ για ένα λεπτό. Ε, ευχαριστώ για να διατηρήσει την εξουσία ε, που είναι στην οποία είναι επιτρέπει τη βία καταστολή ο Λουκασέγκο οποιασδήποτε δραστηριότητα αντιπολίτευση, ακόμα και των δημοσιογράφων που προασπίζονται τα ανθρώπινα δικαιώματα, τα μενοτικά δικαιώματα, ή αυτών που ε, ασκούν ελεύθερο συνδικαλισμό. Υπάρχουν και άλλοι. Ο κύριο Σεμπελίτσκι, παραδείγματο χάρη, του Κέντρου Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τη Βιάσνα, ο οποίο συνελήφθη. Και αυτό είναι δείγμα αυτή τη καταστολή και θα πρέπει να απελευθερωθεί και ο ίδιο και όλοι οι άλλοι κρατούμενοι που κρατούνται γιατί ε, αντιτάχθηκαν στο καθεστώ. Το κοινοβούλιο μα θα πρέπει να ζητά επίση να ζητήσει μορατόριο των εκτελέσεων ε, και πλήρη κατάργηση τη αντική ποινή. Το διεθνέ εμπορικό κίνημα θα πρέπει να δείξει έμπρακτα τη στήριξή του στους Λευκορώσους, θα πρέπει ε, τα συνδικάτα να ε, λειτουργήσουν και να καταγγείλουν ε, τις ιδιωτικοποιήσεις, τον έλεγχο των τροφίμων και να φροντίσουν ο πλούτος να χρησιμοποιείται προς όφελος των πολλών και όχι της μικρής οικονομικής και πολιτικής ελίτ. Ευχαριστώ κύριε Μέρφη. Ο κύριος Πάσκα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Ε, κύριε Πρόεδρε, κύριε Επίτροπε. Καμιά φορά στον κόσμο οι ηγέτες που δεν χαίρουν ε, τη υποστήριξη του πληθυσμού να ψάχνουν τρόπο να κρατηθούν στην εξουσία. Όσο περισσότερο θέλει ο λαός να απελευθερωθεί από αυτό το δυνάστη, τόσο πιο ε, σκληρές μεθόδους χρησιμοποιεί κατά της κοινή γνώμης αυτός. Οι δημοσιογράφοι και οι επικριτικοί πολίτες είναι οι πρώτοι που υφίστανται τα αντίπεινα και είναι εκείνοι που εκφράζουν εκείνους που θέλουν την πολιτική αλλαγή στη χώρα. Η κυβέρνηση έχει θορυβηθεί και ανησυχήσει για τις επόμενες βουλευτικές εκλογές ε, στη Λευκορωσία διότι η κοινή γνώμη όλο και περισσότερο αφίσταται και απομακρύνεται από το καθεστώς οι πιστοί του Λουκασέγκο επιβραβεύονται για τη δουλειά τους, αλλά η αλλαγή θα μπορούσε να σημάνει ε, απώλεια των προνομίων τους. Γι' αυτό δεν διστάζουν να ε, κακοποιούν τον ποινικό κώδικα, να εκφοβίζουν ε, τους πολιτικούς αντιπάλους και τους δημοσιογράφους. Η συνεδρίαση των Υπουργών Εξωτερικών των χωρών της ε, Ανατολικής Γειτονίας είναι μια καλή ευκαιρία να διατρανώσουμε στους Λευκορώσους ότι όλα αυτά είναι απαράδεκτα. Ευχαριστώ κύριε Πάσκα. Αυτοί ήταν οι ομιλητέ εξ ονόματο των πολιτικών ομάδων και τώρα η υπόλοιποι, η κυρία Γιάκον Σάρη, για ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, συνάντησα τους πολιτικούς κρατούμενους ε, στην Λευκορωσία Συνήθω ήταν δημοσιογράφοι, όπω στη συγκεκριμένη περίπτωση συναντήθηκα με συνδικαλιστέ, ακτιβιστέ και πολλά μέλη κομμάτων που έχουν φυλακιστεί. Πολιτικοί φυλακισμένοι δεν θα έπρεπε να κρατούν, δεν θα έπρεπε να υπάρχουν. Αλλά η κατάσταση στην Λευκορωσία σε ό,τι φορά τα ανθρώπινα δικαιώματα επιδεινώνεται μέρα με τη μέρα. Γι' αυτό τον λόγο η δράση τη Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να είναι πιο ενεργή, πιο, να είμαστε πιο δραστήριοι να παρακολουθούμε εκ του σύνεγγυς εξελίξεις και να επεμβαίνουμε. Αυτό είναι ακόμα πιο σημαντικό, πολλό δε μάλλον τώρα που προετοιμάζεται η συνάντηση των Υπουργών Εξωτερικών. Σε αυτό το πλαίσιο, σε αυτή τη συνάντηση, χρειάζεται να θίξουμε το ζήτημα της επιδείνωσης των δικαιωμάτων στη Λευκορωσία. Πρέπει να δώσουμε μεγαλύτερη στήριξη προς τους νέους, τους φοιτητές που επιθυμούν να ταξιδέψουν και να σπουδάσουν στην Ευρώπη. Ευχαριστώ πολύ κύριε Γιακονσάρη. Κάτσε διάει. Και εδώ έχω πολύ περισσότερους από όσους μπορώ να δώσω το λόγο. Παρακαλώ να δείξετε κατανόηση. Θα δώσω το λόγο σε εκείνους που δεν μίλησαν προηγουμένως. Και όχι σε όλους. Ο συνάδελφος Πρωτασίεβιτς. Ευχαριστώ πολύ, panie przewodniczący. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Προεβδομάδος όταν προτάθηκε το ψήφισμα ο κύριος Ποτσοβούτ βρισκόταν ακόμα στη φυλακή. Τώρα αποφυλακίστηκε. Θα ήθελα να πω μερικά λόγια για τον κύριο Ποτσοβούτ διότι τυχαίνει να τον γνωρίζω προσωπικά. Ήρθε να με επισκεφθεί στην Πολωνία είναι ένας πραγματικά ακέραιος άνθρωπος και ε, κάνει πολύ καλή δουλειά στην Λευκορωσία ως ε, μέλος ε, συνδικάτου. να αναφέρω το όνομα του Άντα Μίχνιχ ο οποίος αντιμετώπισε παρόμοιες καταστάσεις. Η Λευκορωσία έχει να χάσει εάν ε, χάσει τον ε, Ποτσκομπούτ. Θα πρέπει λοιπόν το καθεστώς να παραπάψει να διώκει άτομα σαν τον Ποτσκομπούτ. Ευχαριστώ κύριος Λίσεκ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πολλοί είναι αυτοί που λένε πάλι ψήφισμα για τη Λευκορωσία. Μα δεν έχει καμία, ε, καμία αξία, δεν τον νοιάζει το Λουκασέγκο. Ίσως όμως, ίσως λέω, τα μηνύματα που εκπέμπουν προς τη Λευκορωσία λαμβάνονται, είμαι βέβαιος εγώ προσωπικά ότι λαμβάνονται από τη Λευκορωσία. Υπάρχει μια ομάδα ε, ανθρώπων γύρω από τον Λουκασέγκο που απολύουν άτομα από τις θέσεις τους είτε γιατί εργάζονται στην αντιπολίτευση, είτε γιατί ε, αγωνίζονται υπέρ της ελευθερίας έκφρασης. Διώκονται μέχρι και φοιτητέ από τα πανεπιστήμια. Θα τους θυμόμαστε αυτούς και δεν θα έρθουν ε, στην ε, Ισπανία να κάνουν ε, τα μπάνια τους, ούτε θα έρθουν στα βουνά μας να κάνουν σκι. Θα τους θυμόμαστε και εμείς. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Λίσεκ. Η κυρία Σαΐα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Η Λευκορωσία συχνά πυκνά επανέρχεται στις εργασίες μας είναι ένα καταπιστικό καθεστώς, αλλά αυτή τη φορά η παραβίαση αφορά έναν Πολωνό ε, δημοσιογράφο που προσωπεί την πολωνική μειονότητα. Ακόμα και αν απελευθερώθηκε, διαπιστώσαμε επανειλημμένα στο παρελθόν ότι οι ποινές δεν ε, ακυρώθηκαν. Στο παρελθόν είχε ήδη καταδικαστεί για αδικήματα εντός εγωγικών τα οποία έχει διαπράξει. Ε, γνωρίζουμε ότι υπάρχουν και άλλοι πολιτικοί κρατούμενοι στις ε, φυλακές. Εγώ υιοθέτησα έναν πολιτικό κρατούμενο στην Λευκορωσία, ο οποίος βασανίστηκε και κάνω έκκληση προς την Κομισιόν ώστε οι πολιτικοί κρατούμενοι να, α, να απελευθερωθούν άμεσα. Ευχαριστώ κύριε Χολμάγερ. Συγγνώμη κύριε Σόμπερμαϊ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Μαζί με το δημοσιογράφο ε, Πάτσο το θέμα της ελευθερίας του τύπου. Ωραία τι χαρακτηρίζουμε τέταρτη εξουσία στην Ευρώπη. Είναι πάρα πολύ σημαντικό στοιχείο της δημοκρατίας. Βέβαια, πώς μέχρι ποιο βαθμό μπορεί κανείς να εξυβρίζει ε, από τα μέσα ενημέρωσης. Είναι πολύ δύσκολη μετάβαση από μια κομμουνιστική δικτατορία στη δημοκρατία. Αλλά είναι υπερβολική η ποινή που έχει επιβληθεί στο δημοσιογράφο. Καταλαβαίνω την αντίδραση ορισμένων Ευρωπαίων πολιτών. Είναι πολύ της ο κύριος Πότσομπουτ, εργάζεται και ζει εκεί ε, στην Ευρώπη θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ ε, ευαίσθητοι ε, στην ανάμειξη στα εσωτερικά μιας χώρας και στον αποκλεισμό της χώρας από το ευρωπαϊκό γίγνεσθε. Αυτός είναι λάθος τρόπος. Και όταν πρόκειται για ελευθερία της έκφρασης και ελευθεροτυπία δεν θα πρέπει να έχουμε δύο μέτρα και δύο σταθμά. Όταν έχουμε σημαντικούς εμπορικούς εταίρους από την Άπο μέχρι την Αραβική Χερσόνησο κάνουμε τα στραβά μάτια. Ευχαριστώ κύριε Όμπερμαγερ. Ε, δέχεστε μια ενδιάμεση ερώτηση του κυρίου Μιγκάλσκι. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Μια σύντομη ερώτηση. Εσείς υποστηρίζετε τη φυλάκιση του κυρίου Πότσομπουτ ή όχι. Ή θεωρείτε ότι είναι ένα εσωτερικό ζήτημα της Λευκορωσίας και να μην ανακατευτούμε. Ή είναι δουλειά μας να το κάνουμε. Δεν το κατάλαβα πάρα πολύ. Ε, ε, εσείς γι' αυτό πληρώνεστε, για να καταπολεμάτε ε, τύπους ε, και συμπεριφορές τέτοιου είδους. Ευχαριστώ απάντηση ε, κύριε Μικάλσκι για την ερώτηση. Μου δίνετε την ευκαιρία να διευκρινίσω γιατί σε ένα λεπτό μέσα δεν μπορούσα να τα πω. Βεβαίως είναι μια ευκαιρία και είναι και ένα θέμα των ευρωβουλευτών να ε, αποφανθούν, αλλά θα πρέπει να είμαστε ισορροπημένοι στον τρόπο με τον οποίο μετρούμε και αξιολογούμε τις ε, παραβιάσεις. Γιατί σε κάποιες άλλες χώρες που είναι λίγο μεγαλύτερες και λίγο σημαντικότερες από τη Λευκορωσία, είμαστε πιο ανεκτικοί. Και βεβαίως θα πρέπει στο διάλογο να υποστηρίξουμε τη Λευκορωσία στη δύσκολη μετάβαση στη δημοκρατία, αλλά είμαστε και πάρα πολύ ευαίσθητοι και να μην ξεχνούμε ότι βεβαίω θα πρέπει να ασχολούμαστε με εκείνου που απειλούνται. Είναι πολύ λεπτό το θέμα. Ευχαριστώ κύριε Ομπερμάγερ. Η κυρία κολασκα Μπομπίνσκα. Ε, ε, Ευχαριστώ πολύ. Στη διάρκεια των συναντήσεων της Ανατολής Ιταλικής Σχέσης, οι εκπρόσωποι της Λευκορωσίας ε, έλεγαν και συνεχίζουν να λένε ότι ε, παραμερίζεται η Λευκορωσία, ουσιαστικά δεν έχει την σωστή μεταχείριση, ενώ ταυτόχρονα συνεχίζει η χώρα την αντιδημοκρατική της ε, συμπεριφορά, ρίχνοντας ανθρώπους φυλακές και αγνοώντας ε, συνεχώς τα μηνύματα τα οποία συνεχώς τις στέλνουμε. Καλό λοιπόν την Ανατολική Εταιρική Σχέση τους Υπουργούς Εξωτερικών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης να επανεξετάσουν τις σχέσεις με τη Λευκορωσία. Λαμβάνοντας υπόψη το ότι συνεχίζει να αγνοεί αυτά που λέμε η Λευκορωσία και συνεχίζει να παραβιάζει ανθρώπινα δικαιώματα. Η Λευκορωσία πρέπει να κατανοήσει αυτά που της λέμε. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Κολάρσκα Μπομπίνσκα. Η κυρία Τούνεν είναι τελευταία. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Χθε ε, ήταν που απορρίψαμε την άκτα, διότι κάποια θέματα δεν είχαν ακόμα σαφή, δεν είχαν αποσαφινιστεί. Εμείς ε, ε δεν θέλαμε να περιοριστεί η χρήση το διαδικτύο. Ήταν δύσκολη η απόφαση την οποία λάβαμε, αλλά τα καταφέραμε, διότι η ελευθερία της πληροφόρησης είναι θέμα πολύ σημαντικό για μας. Και σήμερα ζητάμε από την Λευκορωσία να εφαρμόσει κάτι το παρόμοιο. Αυτό το οποίο πράττουν μέχρι τώρα οι αρχές της χώρας είναι απαράδεκτο. Μέλη της δημοκρατικής ε, αντιπολίτευσης ε, όπως ο Πόσκο Μπούντ ε, θα πρέπει να τύχουν τη στήριξη των ευρωπαϊκών θεσμικών οργάνων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία τον Χόσταν. Προκρίνονται και η διαδικασία ΚΑΤΣΙΑΗ και η Επίτροπος έχει το λόγο. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Στις 23 Σεπτεμβρίου η Λευκορωσία έχει βουλευτικές εκλογές και η συζήτηση αυτή είναι πάρα πολύ επίκαιρη. Γνωρίζουμε όλοι ότι η ελευθερία της έκφρασης είναι θεμελιώδη στοιχείο για οποιαδήποτε ελεύθερη προεκλογική εκστρατεία. Και είναι πάρα πολύ σημαντικό να στείλουμε αυτό το τόσο ισχυρό μήνυμα από ένα ευρύ φάσμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είπα ότι εκπρόσωπο Άστον ανησυχεί βαθύτατα και παραμένει ανήσυχη για τι κατάφορε παραβιάσει ανθρωπίνων δικαιωμάτων, κράτου δικαίου και δημοκρατικών αρχών στη Λευκορωσία. Από τον Απρίλιο όταν Σάνικο και Παρανταρένκα αφέθηκαν ελεύθεροι, επιφανεί πολιτικοί κρατούμενοι, δεν υπήρξε καμία άλλη απελευθέρωση πολιτικών κρατουμένων. Και εκείνοι που έχουν αφαιθεί ελεύθεροι υφίστανται τεράστιους περιορισμούς στα πολιτικά τους και αστικά δικαιώματα. Σε αντίθεση με αυτό, ε, είδαμε ε, μεγαλύτερη καταστολή ε, των δημοσιογράφων, των μέσων ενημέρωσης με διοικητικά πρόστιμα και επιβολή κυρώσεων και ποινών. Την περασμένη εβδομάδα ο εκπρόσωπος της κυρίας Άστον εξέφρασε τη βαθιά του ανησυχία για τα όσα μαθαίνουμε για παρενόχληση εκπροσώπων της κοινωνίας των πολιτών, της αντιπολίτευσης και ε, ανεξαρτήτων μέσων ενημέρωσης. Η ελευθεροτυπία παραμένει ε, σε καταστολή και σε μεγάλο βαθμό και η ανεξάρτητη δημοσιογράφη συχνά είναι στόχος ε, των αρχών. Ο εκπρόσωπος της κυρίας Άστον έκανε ιδιαίτερη αναφορά στο δημοσιογράφο Ανδρέη Πότσοβουτ που ακριβώς ε, ασκώντας ε, το λειτουργήμα του δημοσιογράφου και για ε, αυτό το λόγο διώχθηκε για συκοφάντηση του Προέδρου. Τον άφησαν ελεύθερο στις αρχές της εβδομάδες αλλά δεν έχουν αποσύρει τις κατηγορίες που του είχαν απαγγελθεί. Και άλλες περιπτώσεις είναι η καταδίκη του Πάιβαλ Σιάρκοφ σε 15 ε, μέρες διοικητικής κράτησης επειδή δήθεν ε, προέβησε δημόσια εξύβριση. Προετοιμάζεται για τις εκλογές του Σεπτεμβρίου η χώρα και επικρατεί γενικά ένας φόβος ε, η ελεύθερη ανεξάρτητη πολιτική δήλωση ή εκδήλωση δεν γίνεται ανοιχτή και οι ανεξάρτητοι δημοσιογράφοι συστηματικά δεν αφήνονται, εμποδίζονται να ασκήσουν τις δραστηριότητε τους. Γι' αυτό είπα ότι εκπρόσωπος και πάλι καλεί τις αρχές της Λευκορωσίας να σταματήσουν κάθε είδους παρενόχληση εκπροσώπων ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης, κοινωνίας των πολιτών και της πολιτικής αντιπολίτευσης και να αντιστρέψουν τη σημερινή πολιτική καταστολή για την κυρία Ισαΐα και άλλους που ζητούν ε, αύξηση των προσπαθειών πρέπει να πω ότι έχω νέα να σας δώσω. Από σήμερα έχουμε μια νέα εξέλιξη. Το Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ ε, σήμερα ε, το πρωί ενέκρινε ένα ψήφισμα που είχε καταθέσει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την κατάσταση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. 22 ναι 20 αποχές και 3 ψήφοι κατά. Το ψήφισμα αυτό ε, απευθύνει επίγουσα έκκληση στην αρχή της Λευκορωσίας να αφήσει ανεφόρον και αμελητή όλους τους πολιτικούς ε, κρατούμενους ελεύθερους και να τους αποκαταστήσει. Και επίσης ορίζει το ψήφισμα ε, το διορισμό ειδικού ε, εισηγητή για τη Λευκορωσία που σε αιτήσια βάση θα αναφέρει στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και στη Γενική Συνέλευση των Ηνωμένων Εθνών. Πιστεύω ότι αυτό είναι μεγάλη επιτυχία της Ευρωπαϊκής Ένωσης που αυτή τη φορά εκέρδισε πολλές ψήφους υπέρ και λίγες ε, κατά ακριβώς για το διορισμό ειδικού εισηγητή. Η κατάσταση λοιπόν είναι ε, σοβαρή, αλλά ε, σας έχω και καλές ειδήσει. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Επίτροπε. Έχω λάβει έξι ψηφίσματα. Ολοκληρώνεται εδώ η συζήτηση γι' αυτό και η ψηφοφορία θα γίνει μετά την επόμενη συζήτηση, η οποία αφορά το σκάνδαλο